Okay, colleagues, if everybody, if everybody could take the... Παρακαλώ, καθίστε. Παρακαλώ, καθίστε. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες. And we're going to start in a minute. Σε ένα λεπτό θα αρχίσουμε. Well, can, can we try test for... Σας παρακαλώ, ας κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Μια δοκιμαστική παρακαλώ για να δούμε ότι λειτουργούν τα μηχανήματά μας. Παρακαλώ καθίστε. Παρακαλώ καθίστε. Και σας παρακαλώ, παρακαλώ τα μέλη να ψηφίσουν. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία, κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να ελέγξουμε αν λειτουργούν τα μηχανήματά μας. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι πέρας και θαυμάσια λειτουργούν τα μηχανήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Οπότε, παρακαλώ καθίστε όλοι. Λοιπόν, σας παρακαλώ καθίστε. Έχουμε κοινή συνεδρίαση, όχι μόνο λοιπόν της Επιτροπής Ανάπτυξης, Ελπίζω να υπάρχουν αρκετά καθίσματα για τους προσκεκλημένους μας από την Επιτροπή Γυναικών, τους οποίους ε, θερμά καλωσορίζουμε. Θα σας ε, αφήσω λίγο χρόνο για να καθίσετε. Παρακαλώ. Ναι, τους παρακαλώ, έλα στο Προεδρείο. Όλα τα μέλη έχουν θέση, έχουν κάθισμα. Παρακαλώ το προσωπικό μας να φροντίσει ούτως ώστε να μπορέσουν να ψηφίσουν όλα τα μέλη. Have all members now... Παρακαλώ, ε, έχουν όλα τα μέλη ένα κάθισμα για να μπορούν να ψηφίσουν. Όχι, παρακαλώ το προσωπικό να φροντίσει ούτω ώστε όλοι να μπορέσουν να ψηφίσουν. Okay, we can maybe make sure that... Λοιπόν, λοιπόν, Ωραία, να κρατήσουμε και μερικέ θέσει αν έρθει κανεί ακόμη. Λοιπόν, έχετε όλοι θέση και μηχάνημα, αρχίζουμε την πληροφορία. Έχουμε λοιπόν κοινή ψηφοφορία με την Επιτροπή Γυναικών. Δεν έχω ανακοινώσει. Λοιπόν, περνάμε στο σημείο 13 στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής Ανάπτυξης. Λοιπόν, είναι μια ψηφοφορία για την εφαρμογή του κοινού εγγράφου εργασία του προσωπικού. Είναι το πρόγραμμα δράση για την ισότητα φιλεγό και η κυρία Σουίκα. Είμαστε συν εισηγήτριες από πλευρά των δύο επιτροπών. Κυρία Σουίκα, α, δεν βλέπω, πού έχετε πάει. Α, εκεί είστε, μάλιστα. Θέλετε να πάρετε το λόγο πριν ε, αρχίσει η ψηφοφορία. Όχι, ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που έλαβαν ψηφοφορια οχι ωραια λοιπον θελω να ευχαριστησω ολου του συναδελφου που ελαβαν μερος ε, στην προσπάθεια επίτευξη συμβασμών. Δεν επιτύχαμε σε όλες αυτές τις απόπειρες, αλλά σε πολλέ και ευχαριστώ πολύ και το προσωπικό που εργάστηκε σκληρά για το θέμα αυτό. Λοιπόν, να αρχίσουμε τώρα την ψηφοφορία. Λοιπόν, τροπολογία 49 υπέρ, κατά, αποχές, θα την ελέγξουμε. Θα την ελέγξουμε γιατί δεν ξέρω τώρα πώ διαμορφώνεται η πλειοψηφία. συγγνώμη, Άρχισε η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Εγκρίνεται. Οπότε, τροπολογία 48 υπέρ παρακαλώ. Συγγνώμη, κάναμε λάθος. Ψηφίζουμε τελικά την 50. Οι υπόλοιπε Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 63. άρχιτε ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε. Α, με συγχωρείτε. Έπρεπε να καταπέσει εφόσον εγκρίθηκε η συμβαστική 3. Α, με συγχωρείτε. Άρα καταπέσει. Περνάμε στα 68. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά απο, αποχές να ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίπτεται ε, ναι όχι απορρίπτεται σαφώς σαφώς συγγνώμη συμβαστική 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε. 94. Ψηφίσατε όλοι. Πέρασε. Εγκρίνεται. Κατά τμήματα για την 95. Πόσα τμήματα? Α, περνά και από την άλλη μεριά της σελίδας. Ε, τέσσερα τμήματα. Το πρώτο, υπέρ. Κατά αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο, υπέρ. Κατά Ελέγχουμε το δεύτερο τμήμα, άρχεται η ψηφοφορία. Το δεύτερο της 95. 95 δεύτερο τμήμα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα. Πέρας. Εγκρίνεται. Τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές. Να ελέγξουμε και το τέταρτο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 97 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Α, με συγχωρείτε, πήδηξα μια συμβαστική. Λοιπόν, να επανέλθουμε στη συμβαστική 3Y. Είναι αμέσως πριν την 97. Υπέρ παρακαλώ τη συμβαστική 3 3Y. Υπέρ, κατά. Να την ελέγξουμε. Τη συμβαστική YYY. 3Y, 3Y. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας, εγκρίνεται. Συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, την 97 την ψηφίσαμε, 98 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 99. Υπέρ. Συγγνώμη. Ε, λοιπόν, να δω τι κάνει το L. 99 ποιοι είναι υπέρ, παρακαλώ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 4Y. Ίσως να πρέπει να γίνει εκ νέου αρρύθμιση των ε, συμβαστικών γιατί αλλιώς Λοιπόν, 4Y. Δεν θα εξηγήσω τώρα, δεν θα ζητήσω τον να μας εξηγήσει γιατί 4Y, δηλαδή στα αγγλικά Y, Y, Y, Y, Y. Λοιπόν, παρακαλώ, ποιοι είναι υπέρ αυτή της συμβαστικής κατά αποχές να την ελέγξουμε. Να την ελέγξουμε. Ελέγχουμε τη συμβαστική 4Y. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Σημαστική 7 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Α, έχουμε κατά τμήματα στην 115. Πρώτο τμήμα, παρακαλώ. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά. Λοιπόν, θα ελέγξουμε το δεύτερο της 115. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι μου. Πέρας. Εγκρίνεται. Λοιπόν, 117 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά αποχές... Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Ε, Συμβαστική 23. 23, συμβαστική υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 120 υπέρ κατά αποχές ελέγχουμε την 120 άρχεται ψηφίσατε όλοι στην 120 πέρας απορρίπτεται 122 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 129 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 130 κατά τμήματα διάφορα τμήματα Α, όχι, μόνο δύο. Μόνο δύο. Πρώτο τμήμα τη 130 υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Το δεύτερο τη 130. Άρχιχο. Πέρας. Εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε. Την 131. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας. Απορρίπτεται. Ισοψηφία. 132 υπέρ. Α, α, με συγχωρείτε, έχει είναι δύο τμήματα 132 υπέρ του πρώτου λοιπόν. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 132 υπέρ. Θα ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα της 132 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 138 υπέρ, κατά αποχές. Ελέγχουμε την 138 άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Με το 43 υπέρ. Κατά αποχές. Ελέγχουμε την 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 144 υπέρ. Κατά ε, να ελέγξουμε. Την 144 άρχεται. Ελέγχουμε αν υπάρχουν ε, διαφορετικές απόψεις μεταξύ των μεγάλων πολιτικών ομάδων. Πέρα συγκρίνεται. 140 υπέρ. Κατά αποχέ απορρίπτεται. 146 υπέρ. Κατά αποχέ, απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά εποχέ εγκρίνεται. 149, δύο τμήματα υπέρ, υπέρ του πρώτου. Κατά εποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 149 θα το ελέγξουμε. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 152 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Λοιπόν, 159 υπέρ κατά αποχές θα την ελέγξουμε. Θα την ελέγξουμε άρχιτε. Πέρας απορρίπτεται. 165 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά αποχές, ελέγχουμε την 166. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 164 υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Συμβαστική 11 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 167 υπέρ. Ελέγχουμε την 167. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά να ελέγξουμε και την 168 άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. 172 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 179 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 185 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται σημαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 184 υπέρ κατά θα την ελέγξουμε την 184 άρχεται ψηφίσατε όλοι εγκρίνεται Ω, Κριστιαν, εγκρίνεται. Γι' αυτό ελέγχουμε. 188. Υπέρ κατά αποχές. 188 σήκω και στο χέρι. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 190. Είναι προφορική τροπολογία. Είναι προφορική τροπολογία. Την έχετε εκεί. Ποιοι είναι υπέρ της 190 ε, με την προφορική τροπολόγηση, υπέρ κατά, θα το ελέγξουμε. Ελέγχουμε την 190. Κανείς δεν εξέφρασε αντίρρηση. Αν έχετε αντίρρηση στην προφορική τροπολογία, παρακαλώ να το πείτε. Έχει κανείς αντίρρηση? Έχει κανείς αντίρρηση? Όχι. Όχι. Κοιτάξτε. Οι συντονιστέ δεν εξέφρασαν αντίρρηση. Ας την ψηφίσουμε. Α, υπάρχει αντίρρηση. Ε, ναι, είμαστε κατά ως ε, ομάδα του ΕΛΚ. Έχει κλείσει το μικρόφωνο της Προέδρου. Mm. Αν έχετε αντιρρήσεις, είναι στον κατάλογο ψηφοφοριών, παρακαλώ πείτε μας ότι έχετε αντιρρήσεις για να μην ψηφίζουμε. 190 χωρίς την προφορική τροπολόγηση. Έτσι αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ, χωρίς την προφορική τροπολόγηση. Τις 190. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά Ωραία, α την ελέγξουμε, α την ελέγξουμε, τελειώνουμε τώρα. Χωρί την προφορική τροπολόγηση. Άρχεται. Πέρας. Χωρίς την προφορική τροπολόγηση, γιατί... Ναι, καλά, εγκρίνεται λοιπόν. Κοιτάξτε, εάν στην Επιτροπή, αν κάποιο έχει αντίρρηση σε προφορική τροπολόγηση ή τροπολογία, τότε δεν μπορεί να υποβληθεί σε ψηφοφορία δεν, ε, εκτός αν έχουν αλλάξει κανόνες, δεν είναι θέμα ε, πλειοψηφιών. Αρκεί να έχει κάποιο αντίρρηση. Ωραία. Τώρα πάμε στην 194. Υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 203 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 13 υπέρ κατά αποχές λοιπόν την ελέγχουμε Καλά, καλά, εγκρίνεται. Όχι, όχι, λάθος, λάθος, συγγνώμη. 204 υπέρ. Θα ελέγξουμε τη 204 έρχεται Ψηφίσατε όλοι, πέρας. Α, ε, απορρίπτεται, απορρίπτεται. Απορρίπτεται, με συγχωρείτε. Δεν είναι σωστά τα νούμερα. 205 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 206 δύο τμήματα. Α, όχι, όχι, όχι, δεν είναι σε δύο τμήματα. Υπάρχει μια προφορική τροπολόγηση του ΕΛΚ. Υπάρχουν αντιρρήσεις? Όχι. Ναι, υπάρχουν. Α, καλώς. Δεν μπορεί να τροπολογηθεί η τροπολογία προφορικά. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 206, όπως αρχικά υπευλήθη υπέρ, παρακαλώ, κατά αποχές. Θα την ελέγξουμε. Θα την ελέγξουμε την 206 χωρίς προφορική τροπολόγηση άρχεται. 206. 206 συνάδελφοι. Χωρίς προφορική τροπολόγηση διότι εκφράστηκαν αντιρρήσεις. Πέρας. Εγκρίνεται. 207 υπέρ. Να ελέγξουμε τη 207 άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 208 υπέρ. Κατά... Θα ελέγξουμε και τη 208. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. πέρα. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά... Αποχές. Να ελέγξω 209. Άρχεται. Ψηφίζονται περα πέρας. Εγκρίνεται. 2-10 υπέρ. Κατά αποχέ. απορρίπτεται. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 2-12 υπέρ. κατα αποχε αποχές εγκρίνεται. 2-13 υπέρ. Κατά αποχε εγκρινεται εγκρίνεται. 2-14 υπέρ. Κατά αποχέ. εγκρίνεται. 2.15 υπέρ κατά ελέγχουμε την 2.15 άρχεται πέρας εγκρίνεται 2.16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ ελέγχουμε τη 2.17 άρχεται πέρας εγκρίνεται Λοιπόν, περνάμε τώρα στι συντολικέ αναφορέ. Ε, τροπολογία 1, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 2, υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 3, υπέρ, κα... να ελέγξουμε την 3, άρχεται. 3, 3, 3, ελέγχουμε την 3, άρχεται, Πέρα. Απορρίπτεται. 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Όχι, είναι ταυτόσιμη με την περασμένη, οπότε εγκρίνεται. Είναι ταυτόσιμες. Πάμε στην τροπολογία 10, υπέρ, κατά, δεν την είδα. Ε, ξανά, με τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι ταυτόσημε οι 9 και 10. Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Εγκρίνονται λοιπόν. 14. συμβιβαστική 14 υπέρ κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχέ εγκρίνεται. 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ ελέγχουμε τη 16 άρχεται ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πάμε στα εκτιμώντας, 22 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. «23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 22 ε, 22 εγκρίθηκε. Όχι. Άρα πρέπει να ψηφίσουμε την 23. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 31 ε, υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 28 υπέρ κατά Ελέγχουμε την 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 34 ε, υπέρ. Κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 32. 32 και 33. Είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά Έλεγχος, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 32 ε, και 33 άρχεται. Τέλος. Αγκρίνεται. 36 υπέρ. Ελέξουμε, ελέγχουμε την 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εγκρίνεται.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 41 δεύτερο τμήμα ψηφίζουμε ψηφίσατε όλοι τέλος εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Πάμε στην, στην ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων, η πρώτο εκτιμώντας υπέρ κατά αποχές, το εκτιμώντας C έχουμε να ψηφίσουμε δρούα. γνωμοδότηση δρούα. Ναι, επιτροπή δρούα. Έχουμε τη γνωμοδότηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Λοιπόν, Κοιτάξτε, τότε ακολουθήστε τον συντονιστή σας γιατί εκείνος έχει τον κατάλογο. Έλκα, ακολουθείτε τον συντονιστή σας. Αν θέλετε βέβαια. Αν δεν έχετε λίστα, ε, τρεις μείνανε, τρεις ψηφοφορίες μείνανε. Four, well, there's a handful of votes to do. Άντε τέσσερις. Yeah, no, let, let's start this vote again. Can we stop, stop voting, close that vote? Can we close that vote? Are we going Λοιπόν, να ε, ε, σταματήσουμε και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λοιπόν, δεν μετράει τώρα. Λοιπόν, ψηφίζουμε επί της νομοδότησης της Υποεπιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. you don't have... Για αυτή την έκθεση. Ελκ, ποιο είναι το πρόβλημα, δεν έχετε κατάλογο ψηφοφορίας. Μάλιστα. Εντάξει. Έχετε όμως συντονιστεί. Εάν θέλετε, μπορείτε να τον ακολουθείτε. Να ξεκινήσουμε πάλι εκτιμώντας C της νομοδότησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται εκτιμώντας E υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται έχουμε λίγες ακόμα 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 21. 21. Ε, ε, Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά για την παράγραφο 21. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Και εγκρίνεται. Και τώρα θα ψηφίσουμε επί της γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Και αυτό γίνεται με ονομαστική κλίση. Άρχεται. Μπορούμε λοιπόν να το ψηφίσουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Και εγκρίνεται με 24 ψήφους ε, με 20 ψήφους υπέρ 24 ψήφους υπέρ με και 5 κατά και 13 αποχές να δώσω το λόγο στην κυρία Σουίκα παρακαλώ συνάδελφοι ησυχία παρακαλώ uh, Ευχαριστώ Λίντα. Όπως ξέρετε ήμασταν ε, εισηγητρίες η Λίντα και εγώ και όπως βλέπετε υπήρξε πολλή σύγχυση και διχασμός, όχι μόνο ανάμεσα σε δύο ομάδες, αλλά και ανάμεσα σε περισσότερες ομάδες, στους φιλελεύθερους, στη θέση του ΕΛΚ. Τώρα, εμείς πήγαμε από πλευρά του ΕΛΚ, αλλά θα χρησιμοποιήσω την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω τον ε, κανόνα 52α για να υποβάλω και την θέση της μειοψηφία. Και να σας πω περί τίνος πρόκειται. Όπως γνωρίζετε, πρόκειται για την πρώτη έκθεση περί της εφαρμογή και διάφορες θετικές τάσεις διαπιστώθηκαν μετά από την πρώτη, το πρώτο έτος λειτουργίας του Gender Plan 2 για το, ε, ε, χρόνια, Τη χρονία 2016 με 2020. Λίντα και εγώ ως εισηγήτριες επιλέξαμε τέσσερις θεματικούς πυλώνες, δηλαδή σωματική και ψυχολογική κυριότητα, πρόθεση κοινωνικών δικαιωμάτων. Συγγνώμη κυρία Σουίκα, κοιτάξτε, εσείς εκεί πίσω κάνετε πολύ φασαρία, πολύ θόρυβο, ε, παρακαλώ ησυχία. Και ακούστε, αν δεν θέλετε να ακούσετε την ομιλήτρια, μπορείτε να φύγετε από την αίθουσα. Ε, λοιπόν, ε, δουλέψαμε επί τεσσάρων αξώνων, θεματικών αξώνων, πρόθεση οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, ε, η χειραφέτηση γυναικών και κοριτσιών, ενίσχυση των, της συμμετοχής στις υπηρεσίες της Κομισιόν, αλλά και στη θεσμική κουλτούρα του τις υπηρεσίε Εξωτερικής Δράσης. Συρίζουμε τις συστάσεις για την περαιτέρω βελτίωση του μέσου. Διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ νωρίς για πλήρη αξιολόγηση του αντικτύπου του ή για επικρίσεις κατά της επιτροπη Επιπλέον είμαι ευεπισμενη ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα πρέπει να εστιάζεται αυστηρά στις πρακτικές πτυχές της εφαρμογη Κατά συνέπεια, δεν μπορώ να υποστήριξω τι τροπολογίε ιδεολογική φύση που ξεπερνούν το πεδίο εφαρμογή και το στόχο αυτή τη έκθεση, τα μη ρεαλιστικά αιτήματα όσον αφορά την αναπτυξιακή συνεργασία τη Ένωση με τρίτε χώρε, καθώ και υπερβολικά δημοσιονομικά αιτήματα, δηλαδή αιτήματα για αύξηση των ε, οικονομικών πόρων, ε, ειδικά όσον αφορά τις αμβλώσεις, ώστε να καλυφθεί το κενό που άφησε η απόσυρση των ΗΠΑ. Να πω λοιπόν και πάλι ότι θα χρησιμοποιήσουμε τον κανόνα 52α και θα υποβάλουμε την μειονοτική μας αυτή θέση ώστε να περιληφθεί σε αυτήν την έκθεση. Ε, σας ευχαριστώ για τη συνεργασία και θέλω να ευχαριστήσω τη Λίντα Μακάβαν που συνεργάστηκε εργαστά μαζί μου, αλλά υπήρχαν κάποιοι συνάδελφοι που, δεν, που είχαν διαφορετικές απόψεις και δεν μπορέσαμε να βρούμε συμβαστικές λύσεις, γι' αυτό και χρησιμοποιώ αυτή την ευκαιρία. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Οποιοδήποτε μέλος έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό ως εισηγητής. Εσείς θα υποβάλλετε στην γραμματεία τη δική σας αυτή γνώμη και θα προσαρτηθεί ε, στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σουίκα για τη συνεργασία. Ευχαριστώ συνάδελφοι. Θα, περάσω, θα αφήσουμε τώρα αυτό το σημείο και θα περάσουμε στο σημείο 14. Σωστά. Η, ε, καλύτερα θα είναι ναι, να αφήσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ώστε να φύγουν οι συνάδελφοι από την Επιτροπή ε, Γυναικών. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία.